ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έλαβε από την ομάδα ΕΛΚ το αίτημα να οριστεί ο κύριος Φράνσις Τζάμι Ντίμεχ ως μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ. Έχει κανείς ε, παρατηρήσει από αυτού? Όχι. Ωραία. Οπότε θεωρείτε ότι εγκρίνεται αυτός ο